Äh, Good afternoon, everyone. Could I call? Um, Καλό απόγευμα σε όλους. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας. Μπορέσαμε να πάρουμε αυτή την επίσημη φωτογραφία με αρκετή αποτελεσματικότητα. Κάποιες σύντομες ε, ανακοινώσεις θα εξετάσουμε σήμερα ένα, ένα εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα για την τεχνητή νοημοσύνη, τα ηθικά ζητήματα που τίθενται και άλλα ζητήματα, αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, μην το ξεχνάμε και αυτό. Σας καλωσορίζω λοιπόν ως αντιπρόεδρος ε, υπεύθυνη για την ε, το διάλογο με τις θρησκευτικέ οργανώσεις αλλά και μη θρησκευτικέ. Καλωσορίζω τους εκπροσώπους της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, ε, Έρευνας και Ενέργειας και τα μέλη του πάνελ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας. Έχετε μπροστά σας ε, ένα, μια σειρά από έγγραφα που θα είναι χρήσιμες και για σήμερα αλλά και για τις μελλοντικές συζητήσεις που θα ακολουθήσουν ελπίζω τη σημερινή. Υπάρχει στη διερμηνία γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, τσεχικά και ελληνικά το σεμινάριο αυτό αναμεταδίδεται ζωντανά. Θα υπάρξει και επίσημος φωτογράφος ε, ε, κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Επίσης, στα μέσα της συνάντησης θα διακόψουμε για καφέ ή τσάι. Καλώς ήρθατε όλοι. Θα βγάλω την, ε, το σακάκι μου γιατί κάνει ζέστη και μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Δεν θα πω πολλά. Ήθελα απλώ να σα πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι τόσοι εμπειρογνώμονε εδώ στα πάνελ μα, αλλά όλου ιδιαίτερω θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Έρευνα ε, Επιστήμη και Καινοτομία, τον Κάρλο Μοέδα, ο οποίο είναι και πολύ καλό φίλο ε, προσωπικό, αλλά και του Κοινοβουλίου. Γενικότερα, γενικότερα είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία τόσα χρόνια και πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα που ήρθατε εδώ, που μα αφιερώνετε το χρόνο σα. Είναι ο δικό σα τομέα πραγματογνωμοσύνη έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό τη τεχνητή νοημοσύνη πολλάκι στο παρελθόν. Εδώ βεβαίω είναι κάπω διαφορετικά τα πράγματα σε αυτή τη συζήτηση, αλλά σίγουρα θα το λάβετε υπόψη σα ε, στην παρουσίασή σα. Καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε, σα καλωσορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σήμερα διότι ο Αντιπρόεδρος Μαγκίνες έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά με βάση τα καθήκοντά της ως υπεύθυνη για τον διάλογο με τις θρησκευτικές οργανώσεις ε, ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλους μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ε, μια παράθεση από κάποιον που μου αρέσει πολύ. Ο Άρτουρ Σι Κλάρκ είχε πει ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει ανώτερη επιστήμη και κατώτερη ηθική, διότι ο συνδυασμός των δύο αυτών είναι αυτοκαταστροφικός. Αυτό έλεγε ο Άρθουρ Σι Κλάρκ. Και όσο πιο πολλά γνωρίζουμε για τον ψηφιακό κόσμο, όσο πιο πολύ μπαίνουμε στον ψηφιακό κόσμο, όλο και πιο σημαντικός είναι ο ρόλος ο δικός μας, ε, όπως ε, εδώ σήμερα, εν πάση Μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε τα πάντα σήμερα, Μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε αριθμούς, ιδέες, αλλά δεν μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε συναισθήματα, εμπειρίες και αυτό κάνουμε εμείς εδώ σήμερα. Ε, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και μέσω Skype. Αλλά δεν μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε τα πάντα. Κάποια πράγματα δεν ψηφιοποιηθούν ποτέ. Και έρχομαι λοιπόν στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης αυτής καθ' αυτής. Διότι δεν πρόκειται για μια τεχνολογία. Ε, πρόκειται για ένα καινούριο κόσμο. Ένα, μια γέφυρα προς ένα καινούριο κόσμο. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον δημιουργό του ίντερνετ, τον κύριο Λί, ε, και πραγματικά μου άνοιξε τα μάτια. Ο άνθρωπος αυτός εφήβρε το διαδίκτυο ε, και ήταν πολύ ε, αισιόδοξο για την επιστήμη τότε και μου είπε στη, συνέχεια ότι αυτός, αυτή η αισιοδοξία έχει πλέον ε, χαθεί επειδή υπάρχουν καταχρήσεις και κάποιοι κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους εκεί, κάποιοι λίγοι. Είπε ότι πρέπει να υπάρχει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για το διαδίκτυο και σκέφτηκα ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και ένα κοινωνικό συμβόλαιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε βέβαια ένα πλεονέκτημα διότι όταν ο κύριος Λί ε, φίβρε το ίντερνετ δεν ήξερε τίποτα για το μέλλον, δεν ήξερε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σήμερα όμως έχουμε μια εμπειρία από τη λειτουργία του ίντερνετ. Εξετάζουμε λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη και μπορούμε να σκεφτούμε τι ακριβώς θέλουμε να εμπεριέχει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τεχνολογικό το ζήτημα. Εγώ είμαι μηχανικός. Συνήθως ε, όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη μιλάμε για τεχνολογικές επιλογές. Όμως η πιο σημαντική επιλογή που έχουμε να κάνουμε δεν έχει να κάνει με την τεχνολογία. Θα ήθελα λοιπόν να πω πρώτα τρία πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην δομή του πώς σκεφτόμαστε το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρώτο έχει να κάνει ακριβώς με την ηθική που μας απασχολεί σήμερα. Με βάση την εμπειρία μου ως μηχανικός ε, και πολλοί συνάδελφοι που εργάζονται στον τεχνολογικό τομέα θεωρούν ότι τα ζητήματα ηθικής είναι ένα εμπόδιο και αυτό πρέπει να σταματήσει. Η ηθική ε, είναι η πηξίδα μας, είναι αυτό που μας διαφοροποιεί και ως Ευρωπαίους, αν θέλετε. Μπορούμε να διαφορο... διαφοροποιήσουμε τον εαυτό μας σήμερα στον κόσμο ε, σε σχέση με το όραμα που έχουμε για το μέλλον. Και το όραμα που έχουμε για το μέλλον είναι διαφορετικό από ό,τι αλλού στον κόσμο. Κάποιοι λοιπόν βλέπουν την ηθική ως ένα εμπόδιο ή το βλέπουν έναν, ως μια, ένας τρόπος να υπάρχουν υπερβολικά πολλές ρυθμίσεις. Και μια από τις μεγάλες εμπειρίες που είχα αυτά τα πέντε χρόνια στην Επιτροπή είναι το πώς ξεφτάσαμε το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Κάποιοι από εμά, ε, πολλοί και στο Κοινοβούλιο, πιστεύαμε ότι τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν μέρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ε, κάποιοι έλεγαν και πάλι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα δημιουργήσει προβλήματα και άλλες ρυθμίσεις και άλλες νομοθεσίες. Δύο χρόνια αργότερα όμως οι άνθρωποι έχουν πλέον καταλάβει ότι είχαμε ένα όραμα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και την προστασία τους. Και αυτό το όραμα ε, γίνεται πραγματικότητα σήμερα. Ε, γίνεται διεθνές πρότυπο. Και εμείς το είχαμε προβλέψει αυτό το 2014 όταν βλέπαμε τα αμερικάνικα κανάλια, όλοι μιλούσαν με άσχημα λόγια ε, για, τα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι το GDPR, μέχρι τη στιγμή που ήρθε εδώ ο, η Apple, ο κύριος ε, Gates και είπαν ότι θέλουμε να κάνουμε το ίδιο με εσά. Κάποια στιγμή έρχονται κάποιοι και μας μιλάνε εμάς πολιτικούς και λένε ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Εάν έχουμε πολλές αρχές, πολλές ηθικές αξίες, ο καθένας θα διαλέγει ε, τη ρύθμιση που τον βολεύει καλύτερα. Θα υπάρχει ένας πληστηριασμός. Θα ψάχνει να περάσει από εκεί όπου δεν υπάρχουν τόσες ρυθμίσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως, διότι το GDPR δεν ήταν έτσι. Διότι έχει σημασία και το μέγεθος. Όταν μιλάμε για 500 εκατομμύρια ανθρώπους που λένε στον κόσμο ότι τα δεδομένα σχετίζονται με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τότε ο κόσμος ακούει. Στις ΗΠΑ υπάρχει αυτό που ονομάζουμε California effect. Όταν δηλαδή στην Καλιφόρνια ψηφίζεται ένα νόμο στη συνέχεια ακολουθούν και, και άλλες πολιτείες, διότι η Καλιφόρνια είναι τόσο ισχυρή οικονομικά, που όταν παράγεται ένα συγκεκριμένο προϊόν, ε, καλό είναι να ακολουθεί την νομοθεσία της Καλιφόρνιας. Νομίζω πως εδώ είχαμε το Brussels effect, δηλαδή την απόφαση αυτή των Βρυξελών προς την προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν δούμε λοιπόν πώς προχωρήσαμε στο θέμα αυτό, το πιο σημαντικό είναι πώς σχεδιάζει την τεχνητή νοημοσύνη και ποιος είναι ο τελικό στόχο. Όταν μιλάμε λοιπόν για το σχεδιασμό, ένα σημείο που για μένα είναι στην καρδιά του ζητήματος είναι η διαφάνεια. Όταν δημιουργούμε τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να γνωρίζουμε τους, αλγο, αλγόριθμους, πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Ιδάλλως δεν υπάρχει διαφάνεια. Είδαμε όλοι ε, αυτό το όχημα στις ΗΠΑ ε, το οποίο ήταν αυτόματο αυτοκίνητο και σκότωσε έναν περαστικό με ένα ε, ποδήλατο, δεν μπορούσε να σταματήσει και τέθηκε το ερώτημα πώς συνέβη αυτό, γιατί το αυτοκίνητο δεν πρόλαβε να δει τον ποδηλάτη και έτσι τον σκότωσε. Όταν όμως δήκανε τον αλγόριθμο, τότε διαπιστώσαμε ότι ο αλγόριθμος εκείνη ακριβώς τη στιγμή αποφάσισε ότι ήταν πιο επικίνδυνο να φρενάρει κάποιος, διότι αυτό ήταν εις βάρος αυτού που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, θα είχε αυτός δηλαδή πρόβλημα, και γι' αυτό δεν φρέναρε. Ήταν απόφαση του αλγόριθμου. Ε, το πιο σημαντικό λοιπόν εδώ είναι να υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι φορά τον αλγόριθμα. αλγόριθμο. Το δεύτερο είναι τα δεδομένα που πρέπει να καλύπτουν όλου του τομεί τη κοινωνία. Πρέπει δηλαδή οριζόντια να καλύπτουν την κοινωνία. Ένα παράδειγμα που δίνω συνήθω είναι κάτι το οποίο όλοι έχουμε ζήσει στην οικογένειά μα. Ένα καρδιακό επεισόδιο. Όταν βλέπουμε τα συμπτώματα, πονάει το αριστερό μπράτσο, σιγά σιγά το στήθος, αυτά είναι συμπτώματα όμως για τους άντρες. Όχι για τις γυναίκες. Γιατί σύμφωνα με την έρευνα, η έρευνα αυτή έγινε με βάση άντρες. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν η ποικιλία όλων των ε, ενδιαφερομένων, τότε δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Όταν λοιπόν προκύπτει ένα τέτοιο ζήτημα με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή θα λειτουργήσει όχι επειδή υπάρχει καλή τεχνολογία, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά και διάφορα δεδομένα τα οποία είναι διαφανή. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς. Το δεύτερο ζήτημα είναι ποιο είναι ο τελικός στόχος. Τι ακριβώ θέλουμε. Μιλάμε με επιστήμονε και του λέμε πότε θα υπάρχει αυτό το ενιαίο σημείο. Πότε η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τόσο έξυπνη ε, όσο οι άνθρωποι. Βεβαίω η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το ίδιο με την ανθρωπίνη νοημοσύνη. Φανταστείτε όμως στο μέλλον κάποιο να αποφασίσει ότι ο στόχος μας είναι να αντικαταστήσουμε τους ανθρώπους. Δεν είναι αυτό το δικό μα όραμα βέβαια. Εγώ θέλω η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει εμένα, να γίνω καλύτερο άνθρωπο, καλύτερο επαγγελματία. Ένα ε, ειδικό για τα θέματα αυτά μου λέει ε, θέλω σε κάποια χρόνια να έχει ο γιατρός μου τεχνητή νοημοσύνη αλλά δεν θέλω να είναι ο ίδιος τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, υπάρχουν μια σειρά από αρχές και εμείς έχουμε εργαστεί σκληρά στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Ηθικής ε, και μπόρεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγώ να προεδρεύσω εκ μέρου του Προέδρου αυτή της, ομάδα, αυτής της ομάδας και αναφέρει το έγγραφο της ομάδας αυτής αυτές τις αρχές. Για να καθορίσουμε λοιπόν ποιο είναι ο τελικός μας στόχος πρέπει να σκεφτούμε τις αρχές μας. Τι θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Θα δεκαταστεί στον άνθρωπο. Όχι. Θα μας κάνει καλύτερους στη δουλειά μας. Πώς θα βοηθήσει τη δημοκρατία τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα βοηθήσει τη βιωσιμότητα. Και τι γίνεται με τη δικαιοσύνη, την ισονομία. Και η μηχανική οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τεχνολογία χρειάζονται οδηγίε, κατευθείαν γραμμέ από ομάδε ε, όπω η δική σα. Βεβαίω υπάρχουν περιοχέ στο, περιοχές στον κόσμο που μπορεί να έχουν διαφορετική μ, μ, γνώμη. Κάποιοι μπορούν να θεωρήσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ελέγχει του ανθρώπου. Δεν είναι αυτή όμω η δική μα βούληση στην Ευρώπη. Καθώς προχωρούμε λοιπόν, πιστεύω ότι το κάθε ζήτημα το οποίο συνδέεται περισσότερο με τις κοινωνικές επιστήμες που συνδέεται με αυτό που κάνετε εσείς εδώ, σε επιστημονικό επίπεδο, σε θρησκευτικό επίπεδο, θα είναι πιο σημαντικό στην ψηφιακή εποχή. Τελειώνοντας λοιπόν θα ήθελα να πω ότι η ηθική είναι μια πράξη αλληλεγγύης και αυτή την αλληλεγγύη την αποδεικνύεται εσείς εδώ σήμερα. Στην Ευρώπη έχουμε δει ποια είναι, τα επιτυχή, ποια είναι η επιτυχία που μπορεί να προκύψει από κοινέ αξίες χωρίς τις οποίες δεν θα ήμασταν σε αυτή την αίθουσα σήμερα όλοι μαζί. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν και αυτού θέλουμε τη συνεισφορά σας, τη συμμετοχή σας για να σχεδιάσουμε αυτήν την τεχνητή νοημοσύνη του μέλλοντος όπου στην Ευρώπη θέλουμε αυτό να γίνει για να βελτιωθεί η ανθρωπότητα, για να έχουμε καλύτερη ζωή, χωρίς όμως να μας αντικαταστήσει εμάς τους ανθρώπους την τεχνητή νοημοσύνη. Ευχαριστώ. Well, thank you, Commissioner. I think you've σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Νομίζω μας δώσατε τροφή για σκέψη και νομίζω ότι όλοι οι συνεπαρόντες εκτιμούν την παρουσία σας. Και κυρίως όσον αφορά τις ε, καταληκτικές σας παρατηρήσεις, πράγματι υπάρχει φόβος ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα υπερκεράσει τον άνθρωπο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια προοπτική και ελπίζω η σύναξή μας εδώ σήμερα να μας προσφέρει αυτή την προοπτική. Ο Επίτροπος ε, θα φύγει, επιτρέψτε μου να τον διευκολύνω, θα λείψω και εγώ για πολύ λίγο και θα παραδώσω την, συντονισμό της συζήτησης στον αδελφό μου, τον κύριο Σβόποντα, που είναι πρόεδρος Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Μπορείτε λοιπόν να διευθύνετε τη συζήτηση για το πρώτο πάνελ.